Ladies Κυρίες και κύριοι, λέω να αρχίσουμε. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω. Γιατί άραγε κάθονται όλοι προς τα πίσω ενώ είναι τόσες πολλές άδειες θέσεις μπροστά. Παρακαλώ τους τελευταίους λοιπόν να έρθουν πιο μπροστά για να καθίσουν στα έδρανα εδώ μπροστά μου. Αλλιώς ο άδειος χώρος θα είναι πολύ φαρδής και δεν χρειάζεται. Κρίμα είναι. Λοιπόν, χαίρομαι που βλέπω τόσο ευρεία συμμετοχή και μάλιστα τόσο αργά το απόγευμα στην τελευταία μέρα εργασιών του Κενοβουλίου πριν από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές. Εδώ έχουμε οργανώσει ένα εργαστήριο σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση για την Εξωτερική Πολιτική του Κοινοβουλίου. Το θέμα, αν δεν απατώμε, είναι ο εξυγχρονισμός των εμπορικών κοαμυντικών μέσων της Ένωσης. Θα ήθελα να σας πω ότι το εργαστήριο αυτό, όπως και τα άλλα, μεταδίδεται από το Ιντρανέτ. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ ευρύ ακροατήριο και τα πρακτικά θα τηρηθούν για το κοινό στο, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως βλέπετε το κοινοβούλιο μας είναι πάρα πολύ διαφανές. Λοιπόν, να σας κάνω την εισήγηση λοιπόν. Πριν από τρία χρόνια ο Επίτροπος Δεχόχτο ήρθε εδώ για την ακρόαση που θα επικύρωνε την, τον διορισμό του τότε μας είχε πει ότι έχει την πρόθεση να βελτιώσει τα, τη λειτουργία των υπαρχών των εργαλείων που διαθέτει η Ένωση για την άμυνα στο εμπόριό της. Αλλά είχε πει ότι όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν μόνον αφού θα έχει υποχωρήσει η κρίση. Δεύτερον, πρόσθεσε, η αποτίμηση που πρέπει να γίνει θα βασίζεται εν ώψη και των αλλαγών που μπορεί να επισυμβούν λόγω των συμπερασμάτων της Δόχας. Επομένως, μπορούμε να αναρωτηθούμε αυτές οι, αυτοί οι όροι, αυτές οι συνθήκες που έθεσε ο Επίτροπος έχουν πληρωθεί ή όχι. Η Κομισιόν πάντως προετοίμασε μια νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση της, εργαλεία, της λειτουργίας των εργαλείων αυτών και εμείς τα μελετήσαμε. Έγινε και μια δημόσια διαβούλευση το φουθινόπορο και παραλήλως η Κομισιόν δημοσίευσε μία εκτεταμένη αξιολόγηση των ισχυόντων για την εμπορική άμυνα της Ένωσης. Το, η νομοθετική πρόταση ετοιμάζεται και θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες, ίσως σε δύο μήνες, ένα-δύο μήνες. Τι μάθαμε. Ο, από τη διαδικασία διαβούλευσης είδαμε ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συμφέροντα και απόψεις μεταξύ των ενδιαφερομένων εξαγωγέων, εισαγωγέων, λιανοπολιτών και ούτω καθεξής. Γενικά, οι αντα... Ό, όσοι συμμετέσχουν στην διαβούλευση αυτή ήταν, τάχθηκαν υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας γενικότερα. Και επίσης από τα, από, από συμπεράσματα που είναι δημόσια φαίνεται ότι θέλουν να συμμετάσχουν περισσότερο οι ενδιαφερόμενοι στην επεξεργασία των νομοθεσιών που τους αφορούν. Άλλες συστάσεις τους ήταν παραδείγματος χάρη περισσότερη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βελτίωση δυνατοτήτων αντιμετώπισης απατών, αντιμετώπιση του θέματος της διπλής ε, τιμής σε ανάλογα με την εσωτερική, την εξωτερική πώληση κλπ. κλπ. Και επίσης τα συνδικάτα ζήτησαν και αυτά να έχουν περισσότερο λόγο και ρόλο να παίξουν. Αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στα έγγραφα μέχρι στιγμή της Κομισιόν. Ακόμα δεν καταλάβαμε αν η πρόταση, η μελλοντική αυτή πρόταση θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα αυτά των ενδιαφερομένων. Ενδιαφέρον θα ήταν να ακούσουμε και να δούμε και τι φρονούν οι αρμόδιοι επίτροποι για όλα αυτά. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως το Κοινοβούλιο κατέληξε ότι καιρός είναι να γίνει κάτι, να γνωμοδοτήσει και εκείνο, να έχει περισσότερη πληροφόρηση για να γνωρίζει καλύτερα τι παίζεται, ώστε όταν έρθει η πρόταση στο Κοινοβούλιο να είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να την αναλύουμε. Τώρα θα σας συστήσω τους καλεσμένους μας. Φρανκ Χοφμάιστερ, αριστερά μου, είναι αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας του Επιτρόπου Ντεχούφτ και αρμόδιος για την ενημέρωση και εξυγχρονισμό των εργαλείων που σας ανέφερα. Θα μας αναφέρει τους στόχους της υπηρεσίας του. Ο Φρανκ Χοφμάιστερ ήταν παλαιά μέλος της ομάδας των εξωτερικών σχέσεων και της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν. Έχει ένα διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και υπήρξε αλέκτορ σε διάφορα πανεπιστήμια στη Χάγη, στο Μάστριχτ, στην Οξφόρδη και στο Ευρωίδρυμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στη Φλωρεντία. Ο πρώτος εμπειρογνώμονας μας θα είναι ο δόκτωρ Φέρμοστ που ανήκει στο Παγκόσμιο Εμπορικό Ίδρυμα της Βέρνης. Έχει θητεία και στη Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες και από το 1995 ασχολείται με τους εξαγωγείς και τις σχέσεις με τον ΠΟΕ και δημοσίευσε πολλά βιβλία για αυτά τα θέματα όπως για τον νόμο εναντίον του ντάμπινγκ της Ένωσης. Μετά είναι ο καθηγητής Ιάκωβος Μπουρζουά ο οποίος έχει και αυτός εκτεταμένη εμπειρία για θέματα που αφορούν το εμπόριο και έχει εκπροσωπήσει πολλούς πελάτες του σε προσφυγές. Έχει εργαστεί και για την Κομισιόν ως κύριος νομικός σύμβουλος για θέματα εξωτερικού εμπορίου και για πολλά χρόνια ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας για το αντι-dumping και της προστασίας κατά των παρανόμων εμπορικών πρακτικών. Αρχίζουμε δίνοντας το λόγο στον κύριο Χοφμάιστερ εξ ονόματος της Κομισιόν. Έχετε τον λόγο για δέκα περίπου λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής μου ζήτησαν να παρουσιάσω σύντομα τα επιχειρήματα και τους στόχους ε, της άσκησης εξυγχρονισμού και θα αρχίσω με μία ερώτηση, απαντώντας μάλλον με τη, ερώτηση που έθεσε ο Πρόεδρος. Εάν εκπληρώθηκαν οι συνθήκες τις οποίες προέβλεψε και οι όροι που προέβλεψε ο Επίτροπος Δικούχτ στην ακρόαση τότε. Η απάντησή μου είναι και ναι και όχι, έτσι και έτσι τότε που είχε αναλάβει την θέση του δεν είχαμε προβλέψει το αδιέξοδο του γύρου της Ντόχα και να τραβήξει τόσο πολύ αυτό το αδιέξοδο. Είχαμε προβάλει μια πρωτοβουλία την οποία, η οποία ελπίζαμε να καρποφορήσει αλλά αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι έχουν κολλήσει πολλά ζητήματα, πολλά θέματα αν και έχουμε υψηλές προσδοκίες για την διευπουργική διάσκεψη του χρόνου στο Μπαλί. Να λυθούν τουλάχιστον μερικά ζητήματα εκεί. Δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει την οικονομική, τα οικονομικά προβλήματα, αλλά έχουμε σημάδια, ορισμένα σημάδια βελτίωσης. Τώρα ποια είναι η λογική την οποία να ακολουθούμε. Από τη σκοπιά των προηγούμενων τριών ετών, οι ενδείξεις, ε, ε, ξέρουμε ότι τα μέσα αυτά εμπορικής άμυνας κατάγονται από το 1999. Είναι δηλαδή μια παλιά ιστορία και το περιβάλλον αλλάζει συνέχεια και γρήγορα. Έχουμε νέους μηχανισμούς αντιπίνων, νέους μηχανισμούς ποινών, κυρώσεων και επίσης η πράσινη βίβλος με τους στόχους της το 2007 απέτυχε. Άρα λοιπόν είναι καιρός τώρα να ξεκινήσουμε τη νέα αυτή άσκηση και ο πρόεδρος Μπαρόσο ζήτησε από τον Επίτροπο κ. Ντεγκούχ να αναλάβει αυτή την ευθύνη, αυτή την υποχρέωση και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπήκε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα και οργανώνεται ή μάλλον συνδιοργανώνεται αυτό το εργαστήρι για ένα περίπλοκο θέμα. Όπως ξέρετε έχει γίνει μια δημόσια ακρόαση μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου φέτος πρώτη, πρώτο, δια, πρώτο συνέδριο, πρώτη διάσκεψη και τα αποτελέσματα είναι διασέσιμα από τον Οκτώβριο με τα συμπεράσματα. Δείχνουμε έτσι ότι η Κομισιόν, η Επιτροπή δείχνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά από τις απαντήσεις που ήρθαν σε μας από τους πολίτες μας, από τους ενδιαφέρομενους πάνω από 3.000 ε, απαντήσεις, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από παραγωγούς, 10% περίπου από εισαγωγής και το υπόλοιπο ποσοστό από δημόσιους φορείς, αρχές, ιδρύματα κλπ. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο αριθμός αυτών απαντήσεων από τα, τις οποίες μπορούμε να συνάγουμε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι βασικοί τομείς που καλυφθούν από αυτή την πρωτοβουλία είναι βασικά 7. Διαφάνεια και προβλεψιμότητα πρέπει να αυξηθεί. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η μάχη κατά των αντιπίνων. Θέλουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την επιβολή των αποφάσεων. Πρέπει να δουλέψουν καλύτερα οι ομάδες που εκτελούν την έρευνα και οι, εκτελεστικές, οι ομάδες που εκτελούν. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και τον μηχανισμό ανασκόπησης και αναθεώρησης μετά την πενταετή περίοδο και βεβαίως υπερο, το, τις υπερορίες υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει μία σειρά αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και τον ΠΟΕ που δείχνουν ότι θα πρέπει να εκλεπτύνουμε αυτούς τους μηχανισμούς ε, της νομολογίας ε, και τις διάφορες εξελίξεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της νομολογίας και της κωδικοποίησης. Θα τονίσω λοιπόν μερικά από, μερικούς από αυτούς τους στόχους. Όσον αφορά τώρα τη διαφάνεια και προβλεψιμότητα, εδώ έχουμε την ιδέα να εισαγάγουμε μία ρήτρα μια χρονική ρήτρα όπου αυτές οι αποστολές ε, παραδείγματο χάρη προϊόντων που βρίσκονται υπό εξέταση να μην μπορούν να εμποδιστούν. Να μην τιμωρήσουμε δηλαδή μία μεταφορά ε, η οποία ήδη είναι καθοδόν ε, και να τιμωρηθεί εκ των προτέρων μέχρι ότι περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και αναλυθεί η προσφυγή, αναλυθεί το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον αυτή η το προβλέψιμο και η διαφάνεια να ενισχυθούν και να επιβληθούν με καλύτερο τρόπο. Το δεύτερο θέμα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της πρακτικής μας. Ε, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα τα οποία μπορούν μόνο οι εμπειρογνώμονες και οι ειδικοί να παρακολουθήσουν. Ας πούμε, όσον αφορά τις ε, δημόσιες ανακοινώσεις ε, θέλουμε να συμπυκνώσουμε και να ενσωματώσουμε ορισμένες τέτοιες ανακοινώσεις σε κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να αυξήσουμε την κατανόηση και την αποτελεσματικότητα των πρακτικών της Κομισιόν. Όπως είπατε και εσείς ότι στο σχεδιασμό των κατευθυντηρίων γραμμών πρέπει να περιλάβουμε και της, ε, την κοινή γνώμη και τις απόψεις που λαμβάνουμε από αυτούς τους ερωτηθέντες. Το χρονοδιάγραμμα επίσης αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών πρέπει να προσδιοριστεί. Το άλλο θέμα το, που, είναι στόχος μας είναι η, χρηματο, τα χρηματοπιστωτικά αντίπεινα. Βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες που αποτελούν στόχο των μέσων άμυνας των μέσων εμπορικής άμυνας υφίστανται αντίπεινα ή πιέσεις και να μην, να μην συνεργαστούν με τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Όταν υπάρξει μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να ε, έχουμε έτοιμη μια ισχυρή και ε, διατεταγμένη αντίδραση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ε, υποθέσεις με δική μας πρωτοβουλία, εξοφίτσιο δηλαδή, όπου θα μπορέσουμε να προφυλάξουμε τους ενάγοντες έτσι ώστε να μην ε, επισημανθούν, να μην μπορούν να αναγνωριστούν από τον εναγόμενο. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία στενότερη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων των, τομέων και της Κομισιόν. Εάν υπάρχει λοιπόν μία περίπτωση ιδίας πρωτοβουλίας, την οποία ξεκινάμε εμείς οι λεπτομέρειες, τις υποθέσεις αυτής πρέπει να προέλθουν από τον τομέα. Ε, για, δεν μπορούμε μόνο εμείς ως Κομισιό να ε, επιτελέσουμε όλο το έργο, αλλά θα βασιστούμε συμπληρωματικά βεβαίως ε, και σε στοιχεία από τον τομέα ή στον οποίο εμπίπτει αυτή η υπόθεση. Και τα, οι λεπτομέρειες όλες πρέπει να καθοριστούν αυτή τη συνεργασία. Το τρίτο σημείο είναι η αποτελεσματικότητα και υλοποίηση, εφαρμογή. Εδώ κοιτάμε ακριβώς ε, πώς μπορούμε να ε, ε, εκμεταλλευτούμε τους κανόνες του ΠΟΕ ΣΥΝ, το λεγόμενο WTO+. ένας, από τέτοιο, ένας τέτοιος μηχανισμός του ΠΟΕ είναι ο κανόνας ε, του, της δασμολογικής ποινής ε, ότι η ποινή που επιβάλλεται ε, μέσω του δασμού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την οικονομική ζημία την οποία έχει υποστεί ο ενάγων από τον εναγόμενο. Και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτός ο κανόνας ε, δεν θα επιβληθεί, δεν θα υπάρχει ρήτρα εξαίρεσης όπου διαπιστώνουμε βαριά παραβίαση ε, και σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχει ακριβώς αυτή η ρήτρα προστασίας ε, του συγκεκριμένου ορίου επιβολής κυρώσεων. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών μας προς αυτή την κατεύθυνση για τη βελτίωση της συνεργασίας κατά τη διάρκεια των ερωτοαπαντήσεων μπορώ να ε, εξηγήσω περισσότερα αλλά όσον αφορά τώρα την βελτιστοποίηση των πρακτικών αναθεώρησης κάθε πολλές φορές ζητείται μια αναθεώρηση, μια ανασκόπηση της κατάστασης, μια έκθεση και πολλές φορές ε, η Κομισιόν δεν είναι ευχαριστημένη με την αναφορά αυτή διότι διαπιστώνει ότι έχουν καταβληθεί δασμοί και εν συνεχεία υποχρεώνεται να καταβάλει τον υστέρων, να δώσει πίσω δηλαδή τους δασμούς αυτούς, ε, καταστάσεις τις οποίες θέλουμε να αποφύγουμε. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να έχουμε περισσότερες διάμεσες εκθέσεις για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε πάντοτε την τρέχουσα κατάσταση και να μην μας προλαβαίνουν τα γεγονότα. Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω Έχω λίγο χρόνο ακόμα. Τώρα, οι λεπτομέρειες της κωδικοποίησης, έχουμε πολλές αποφάσεις, ε, μια νομολογία δηλαδή την οποία θέλουμε να ενσωματώσουμε, κυρίως νομικά θέματα ορισμών Επίσης όσον αφορά το θέμα των δειγμάτων, εδώ θα εφαρμόσουμε μια ε, πιο ταχεία διαδικασία, θα επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ε, αυτές ε, είναι καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζουμε μέσα στο, στις υπηρεσίες μας. Δεν νομίζω να υπάρχουν αντιρρήσεις και να είναι επίμαχες Επίσης, ε, ε, ο στόχος μας όλος ε, είναι βεβαίως, όλοι μας οι στόχοι είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, μέσα στην Κομισιόν έχουμε μία διαδικασία ανάλυσης επιπτώσεων. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η ανάλυση, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία υιοθέτηση μιας πρότασης. Προβλέπουμε στις αρχές του καινούριου χρόνου να είμαστε έτοιμοι να, να έλθουμε ξανά στο σώμα, εδώ, στο Κοινοβούλιο, με την τελική μας πρόταση και πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της αξιότιμης επιτροπής σας και από τη δική σας προεδρία θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή, τη μεταρρύθμιση. Η Κομισιόν ενδιαφέρεται και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην μεταρρύθμιση και στον εσυγχρονισμό. Ευχαριστώ πολύ. in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 ε, ακολουθούν το σύστημα αυτό με τα, τις καλές του πτυχές, για παράδειγμα τους κανόνες W ε, του ε, αλλά και με τις αρνητικές του πτυχές. Για παράδειγμα, έλλειψη ε, διαφάνειας, παρόλο που έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει, έστω και παρά τη θέλησή της, ηγετικό ρόλο, έχει συνέπειες ε, επί των προτάσεων που ε, καταθέτει η Κομισιόν, γιατί αν αυτές οι προτάσεις υιοθετηθούν, είμαι 100% σίγουρος ότι θα ακολουθηθούν και από άλλες χώρες. Μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σχολιάσω αυτά τα επτά θέματα τα οποία εντόπισε η Κομισιόν. Πρώτον, η αύξηση της διαφάνειας. Όπως, καταλαβα... καταλαβαίνετε από αυτά που μόλις είπα, για μένα είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα. Γιατί, γιατί είναι η πιο αδύναμη πτυχή του σημερινού υφιστάμενου συστήματος. Βέβαια, το υφιστάμενο σύστημα έχει βελτιωθεί επανειλημμένως, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι ε, έχει μετατοπιστεί και η εστίαση ε, των μέσων εμπορικής άμυνας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη, γεωγραφική εστίαση, το γεωγραφικό εντοπισμό. Ε, στον προηγούμενο αιώνα είχαμε υποθέσει εναντίον της Ιαπωνίας, της Κορέας, των ΗΠΑ σε κάποιο βαθμό, αλλά όλοι γνωρίζουμε την ότι την τελευταία δεκαετία ο βασικός στόχος ε, των υποθέσεων αυτών, των προσφύγων αυτών και των μέσων μάλλον αυτών είναι η Κίνα και το Βιετνάμ. Ε, είναι, δεν είναι οικονομία της αγοράς ε, και αυτό είναι σημαντικό γιατί σε αυτές τις χώρες το σύστημα είναι πιο αδιαφανές από ό,τι στις χώρες που χαρακτηρίζονται από οικονομία της αγοράς. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τις λεπτομέρειες, αλλά να σας πω δύο λόγια σε περιπτώσεις ε, ε, χωρών που δεν είναι η οικονομία της αγοράς ε, λαμβάνεται το κόστος και τις τιμές αναλογικά με μία οικονομία της αγοράς. από αυτές, ορισμένοι από τους φορείς δίδουν πληροφορίες, αλλά όχι όλοι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις η ε, οι ε, στόχοι, οι επιχειρήσεις στόχοι ε, δεν ξέρουν πώς υπολογίζεται κάθε φορά η τιμή. Αυτό δεν συμβαίνει στη οικονομίες αγορά Συνεπώ, στι χώρε που δεν είναι η οικονομία τη αγορά. η αδιαφάνεια είναι μεγαλύτερη. Ορισμένα, ορισμένα μέτρα αναφέρονται στην έκθεση ή ε, τρεις εβδομάδες για παράδειγμα, η τρεις εβδομαδε για παραδειγμα η συνδεση με κάποια ρήτρα ε, ναύλου, αποστολής μάλλον, δεν θα βελτιωθεί πάρα πολύ πάνω στο σύστημα με αυτή την πρόταση. Γιατί ε, αυτές οι προτάσεις ε, πολύ συχνά πριν την εφαρμογή των δασμών γίνονται γνωστές, διαραίουν. Ε, δεύτερον, αν μια πρόταση ε, για προσωρινά μέτρα ε, διαρρεύσει μερικές εβδομάδες πριν, τότε η πρόταση για μία επαβολή θα πρέπει επίσης να ε, γίνει δημόσια. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα επίσης, ε, να δημοσιεύουμε ένα, μια περίληψη της καταγγελίας ε, μόλις κατα, κατατεθεί και όχι όταν ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής ε, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ και όπως συμβαίνει τώρα. Ε, πολλές φορές έτσι και αλλιώς στις ΗΠΑ ο ίδιος ο καταγγέλων διαρρέει την καταγγελία του αλλά ακόμα και όταν δεν τη διαρρεύσει πολύ συχνά διαρρέεται από τρίτους. Οπότε η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε δύο συστήματα. Έχουμε το επίσημο σύστημα που χαρακτηρίζεται από εμπιστευτικότητα μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία και υπάρχει και το άτυπο ανεπίσημο σύστημα στο οποίο όλοι γνωρίζουν κοινό μυστικό η καταγγελία. Τώρα, η εκθέση στο τέλος ε, ε, της διαδικασίας, αν υπάρξουν αιτήματα, αν υπάρξει τέτοιο αίτημα θα πρέπει όμως να δημοσιεύεται. Ε, οι εκθέσεις επιβεβαίωσης, ε, αυτές οι εκθέσεις θα μπορούσαν ε, επίσης να ε, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους. Αν ε, δοθούν πληροφορίες στην Επιτροπή ε, παρόμοιες πληροφορίες θα μπορούσαν να δοθούν και στους ενδιαφέρομενους. Το ίδιο ισχύει και για, τις, και για την Επιτροπή εναντίον, κατά των επιδοτήσεων. Πολύ συχνά δεν, δίνουν, δεν ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Μετά, καταπολέμηση της, των αντι, αντιπίνων. η αυτεπάγγελτες έρευνες ε, δεν είναι απάντηση. Ε, είναι σωστό ε, και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει εδώ, ιδιαίτερα εδώ, οι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν χώρες που ήδη το κάνουν, για παράδειγμα το Περού, έχουν ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για εναντίον της Κίνας, αλλά αυτή είναι μια διαφορετική κατάσταση, γιατί ο κλάδος ε, είναι κατακαιρματισμένος. Ενώ η ιδέα των αυτεπάγγελτων ερευνών, αν δείτε την ιστορία των συμφωνίων αντι-dumping, ε, είναι να αποτελέσουν ε, απάντηση για κατακαιρματισμένου κλάδους. Η απάντηση Κομισιόν όμως πηγαίνει πιο μακριά, δεν αναφέρεται σε κατακαιρματισμό, εκτό και αν κάνω λάθος. Οπότε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτέ οι έρευνε σε άλλου τομεί και άλλε χώρε σίγουρα θα, θα υποφεληθούν. Τώρα, σε πρόσφατες περιπτώσεις αυτά τα ε, αντίπινα εφαρμόζονται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Και αν υπάρχει αιτιολόγηση, αυτή δεν αποκαλύπτει στους ενδιαφερόμενους. Οπότε, κάποιοι λένε ότι, ο... Ε, ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας ε, φόβου περαιτέρω αντιπίνων. Αυτό είναι καινούριο. Πριν από 10 χρόνια δεν συνέβαινε αυτό. Τρίτο, τρί, τρίτος παράγοντας, αποτελεσματικότητα και εφαρμογή των μέτρων. Η, η ιδέα των αυτεπάγγελτων ερευνών ε, είναι θεμητή, έχει άλλωστε εφαρμοστεί ε, στη, από την Κομισιόν. Η μία εφαρμογή του ε, κανόνα του μικρότερου δασμού είναι επίσης σημαντική ε, σε περιπτώσεις ε, ερευνών εναντίον της, ε, της παράβασης, εναντίον, της παράκαμψης. Η τρίτη περίπτωση όμως, η μη εφαρμογή του κανόνος του μικρότερου δασμού σε περιπτώσεις, υποθέσεις εναντίον, της, εναντίον επιδοτήσεων δεν είναι πάντοτε σωστή ε, ιδιαίτερα όταν μερικές ε, φορές τα αιτήματα που προέρχονται δεν είναι ε, παρκώς θεμελιωμένα. Μετά, η, τα αιτήματα ανα, επανεξέτασης ε, ο συνδυασμός επανεξέτασης στο μέσο και στο τέλος δείχνει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι απαραίτητος, δεν είναι πολύ ε, ε, αναγκαίος, διότι έτσι κι αλλιώς οι ενδιαφέρον μπορούν, να ζητήσουν ενδιάμεση επανεξέταση. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να γίνει αυτό ο συνδυασμός, αλλά δεν είναι απαραίτητος. Και τέλος, το ανέφερε ο κ. Σχοφμάιστερ, η πρόταση για την επιστροφή των δασμών ε, αν δεν παραταθούν τα μέτρα είναι δίκαιη. Αυτά. Θα είμαι στη διάθεσή σας. Thank you. And now, Professor Jacques Bourgeois. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Ζακ Μπουρτζουά, από το Κολέγιο της ε, Ευρώπης. Και πάλι 10 λεπτά. Ladies as Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όπως ε, ανέλησε ο αγαπητός συνάδελφος, είμαστε εδώ, καθήμενοι ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά όχι ακριβώς και στην ίδια πλευρά των επιχειρημάτων. Εγώ ενεργώ ο λίγων ως δικηγόρος και σήμερα υπερασπίζουμε τον κατηγορούμενο, αύριο υπερασπίζουμε το θύμα του τεστίν έχω βρεθεί σε καταστάσεις όπου έχω υπερασπιστεί ή κατηγορήσει και τις δύο πλευρές, είτε τον τομέα, τον οικονομικό, είτε τους εισαγωγής, εξαγωγής. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς σε όλα τα σημεία, το ανέφερε ο κύριος Hofmeister, απλώς θα συμπληρώσω με ορισμένα σημεία τα οποία δεν ανέφερε και ο κύριος Βερμούλς επίσης δεν ανέφερε μερικά. Το πρώτο ζήτημα είναι το πώς ξεκινάνε οι προσφυγές, οι έρευνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δέχεται ε, αιτήματα προσφυγών υψηλού επίπεδου. Ε, πιστεύω ότι είναι το υψηλότερο επίπεδο προσφυγών και αιτημάτων που δέχεται από όλους τους άλλους φορείς. Το πλεονέκτημα είναι ότι μειώνεται πολύ σημαντικά ο κίνδυνος στο τέλος της ε, όλης της υπόθεσης ε, να αναγκαστεί να πει η Κομισιόν ότι δεν επήλθε ζημία, δεν υπάρχει παραβίαση κλπ. Το θέμα είναι ότι εδώ έχει σημασία όχι μόνο η χρονική διάσταση, αλλά και το κόστος από τη στιγμή που ανοίγει ένας φάκελος μέχρι τη στιγμή που κλείνει. Και η αξιολόγηση αυτών των ε, μηχανισμών των μέσων εμπορικής άμυνας έχει ένα κόστος μεταξύ 60 και 100.000 ευρώ ε, ε, είναι το κόστος της προετοιμασίας μιας, κατα... μιας προσφυγής. Όταν προσθέσουμε και το κόστος της έρευνας, της ανάλυσης, της μελέτης, όλης της περίπτωσης κλπ, τότε το κόστος της προσφυγής και της χρήσης αυτών των μέσων εμπορικής άμυνας είναι απαγορευτικός και ιδιαίτερα απαγορευτικός για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ ακριβώς θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της η Κομισιόν. Σε αυτό το ειδικό πρόβλημα. Ίσως μπορεί παραδείγματο χάρη να ε, έχει να δημιουργήσει ένα απλουστευμένο ερωτηματολόγιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή κάτι άλλο που μπορούμε να φανταστούμε. Τώρα, οι αυτεπάγγελτες ε, προσφυγές και η, αυτε, αυτεπάγγελτη έρευνα μια προσφυγής μπορεί να μην είναι πάντοτε πολύ χρήσιμη, ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο ευρωπαϊκός τομέας αντιπροσωπεύεται μόνο από δύο-τρεις εταιρείες. Οπότε δεν, δεν θέλουμε να αποκαλυφθεί στην χώρα εξαγωγής ποιες είναι ακριβώς αυτές οι εταιρείες οι ευρωπαϊκές. Όμως τα αντίπεινα είναι ένα σημαντικό και πραγματικό πρόβλημα. Είχα μία περίπτωση, μία υπόθεση, όπου ο ενδεχόμενα εντάγων μου είπε ότι δεν θα συνεχίσω, δεν θα προχωρήσω στην προσφυγή. Και πήρα αυτή την απόφαση επειδή η χώρα εξαγωγής είχε απειλήσει με αντίπεινα. Χώρα εξαγωγών. Ε, δέχεται λοιπόν η Κομισιόν να μην είναι σε θέση να καλύψει τα νόματα των ευρωπαϊκών εταιριών που εμπλέκονται στην προσφυγή και να μπορούν να, κρυφτούν αυτά τα ονόματα. Αλλά θα πρέπει να δώσει ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα στις εξαγωγικές χώρες. Και ε, σε αυτό υποστηρίζουμε την Κομισιόν. Όσον αφορά τώρα τον κανονισμό του, του, του, της χαμηλότερης επιβολής δασμού, είναι ένας κανόνας του ΠΟΕΣΙΝ, WTO+, και πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτόν. Τώρα θα πρέπει να εφαρμοστεί στις, ε, ε, στους δασμούς ε, κατά της απορρόφησης και κατά της that Παρέκκλησης δεν ξέρω εάν θα, αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν αυτές οι δύο περιπτώσεις και αν αυτός ο κανόνας του κατοφή, του, της οροφής ε, του δασμολογίου, του, του δασμού θα πρέπει να επιβληθεί σε περιπτώσεις ε, επιδοτήσεων ή dumping. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις ε, ε, κυρώσεων για dumping και επιδοτήσεις πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας του ποε συν. Ε, και κύριοι πρέπει να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή. Έχουμε ένα σύστημα όπου η Κομισιόν χρειάζεται τη συνεργασία του τομέα των εξαγωγέων και των εισαγωγέων στη μελέτη ενός φακέλου, στη μελέτη μιας υπόθεσης. Ποιες είναι οι κυρώσεις? Μηδέν. Πρακτικά, από πρακτικής απόψεως μηδέν. Ναι, βέβαια, υπάρχει, υπάρχουν ε, ε, ενδείξεις και αν υπάρχουν, ε, υπάρχει το θέμα της, θέματα παράκαμψης, απορρόφησης κτλ. Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια ε, ταχύτερη, συντομότερη διαδικασία η οποία θα καταλήξει σε επιβολή δασμολογικών ποινών. Αλλά αυτές δεν είναι κυρώσεις και αν συγκρίνουμε την κατάσταση αυτή με, τις, με τις κανόνες ανταγωνισμού θα δείτε ότι οι, ευρωπαϊκές, ε, ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού προβλέπουν, προβλέπουν κυρώσεις ποινές σε περιπτώσεις ε, ε, μη συνεργασίας. Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε και παρόμοιες κυρώσεις σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε εφόσον δεν υπάρχει θέληση συνεργασίας. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ του τομέα ανταγωνισμού και των μέσων εμπορικής άμυνας. Εφόσον συζητάμε για προβλεψιμότητα και διαφάνεια, πιστεύω και σε αυτό το σημείο συμφωνώ με τον συνάδελφό μου κύριο Βερμούλης, και τις προτάσεις της Κομισιόν, θα πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές για ορισμένα ζητήματα και ένα περιθώριο ε, ε, ζημίας ε, μιας χώρας, αλλά ομιλώντας ως, νομι, δικηγόρος, δεν βλέπω πώς η Κομισιόν θα μπορούσε να υιοθετήσει κατευθυντήρες γραμμές ε, για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα συμφέροντα της κοινότητας. Ιδίως τώρα που είμαστε μέσα στο σύστημα το, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως καθορίζει τις ε, εξουσίες ε, η συνθήκη της Λισαβόνας. Τι σημαίνει τώρα το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφέρον σημαίνει ότι πρέπει να επισημαίνουμε ε, τις τα διαδικασίες που οδηγούν σε ντάμπινγκ, σε επιδοτήσεις και επιφέρουν ζημία στην Ένωση. Όμως αυτό το παραγωνίζουμε και αποφασίσαμε ότι δεν θα επιβάλλουμε μέτρα τι, μα τι γίνεται, είναι αυτό συνεπές με αυτά τα οποία ορίζει ε, η, το άρθρο 290 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις be for the act. για τις εξουσίες της Ένωσης. Εδώ μιλάμε για νομοθετικές πράξεις και λέει ότι δεν θα πρέπει να υποκείμασα σε πράξεις εξουσιοδότηση. Και όμως υπάρχει υποχρέωση για τον νομοθέτη να καθορίσει τα στοιχεία που θα πρέπει να μελετήσει η Κομισιόν ή υπό τη διαδικασία επιτροπολογίες για να θεωρηθούν, να ληφθούν υπόψη από την Κομισιόν όταν ε, αναλύει και εξετάζει ποιο είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω, Πρόεδρε, να ε, κρατήθηκα μέσα στα χρονικά όρια που μου ζητήσατε και θα απαντήσω με ευχαρίστηση ερωτήσεις. Πράγματι, ας αρχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση με τους βασικά, βασικούς ενδιαφερόμενους. Αυτά συνηθίζω να κάνω εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις. Business Europe, δηλαδή η συνομοσπονδία των επιχειρήσεων στην Ένωση. Είναι εδώ η κυρία Σέρβετ Γκούντρουν, που είναι αντιπρόεδρος της ομάδας εργασίας για τα εργαλεία του εμπορίου της Business Europe. Ορίστε. Για κάνα δυο λεπτά, έστω πέντε, άντε πέντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία στην Business Europe να λάβει το λόγο σε αυτό το εργαστήριο για την εξυγχρονισμό κτλ. Μου λέει ο τίτλος. Τα TDI δηλαδή τα εργαλεία εμπορικής άμυνας κατά του αθέμητου ανταγωνισμού είναι κάτι που το δέχονται όλα τα μέλη μας. Δεν είναι προστατευτικά, δεν είναι εργαλεία προστατευτισμού, αλλά ούτε εργαλεία για να αναδιαρθρώσουν τις εταιρείες. Αντίθετα, σε ένα κόσμο ανοιχτού εμπορίου και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα λόγω των πολυπλοκότητας των εμπορικών σχέσεων πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός καταπολέμησης του αθέμητου εμπορίου. Και αυτό είναι ο μόνος νόμιμος θεμητός τρόπος για να αμυνθούν οι επιχειρήσεις ώστε να διατηρηθούν οι αρχές του δικαίου. Αυτά συμφωνούν και με τη συμφωνία αντι-dumping που ισχύει σχεδόν παντού και στην Ένωση και που ξεπερνάει κατά πολλά τους κανόνες του ΠΟΕ. ώστε να εξισορροπηθούν τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων. Η Ένωση λοιπόν προσφέρει περισσότερα μονομενός από αυτά τα οποία έχει δεχτεί σε διεθνείς συμβάσεις. Εμείς στη Business Europe πιστεύουμε ότι το ίδιο ισορροπημένο εργαλείο αυτό δεν πρέπει να αποδυναμωθεί στο μέλλον ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου δεν συμβαίνει καμία πρόοδος στον ΠΟΕ, που ήταν η μία από τις δύο συνθήκες που είχε θέσει, όρους που είχε θέσει ο πρόεδρος Μπαρός όταν έλαβε τα καθήκοντά του. Το σύστημά μας είναι λοιπόν σωστό και καλό, αλλά νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Πιστεύουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να εισαχθούν ρήτρες για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού για τα πρώτες ύλες. Επίσης πιστεύουμε ότι όταν υπάρχει στρεβλωμένη πρόσβαση σε αυτές, οι ανταγωνιστές έχουν το πλεονέκτημα μέσω άμεσων ή έμεσων επιχορηγήσεων προς τις εξαγωγές και αυτό καταλήγει πρακτικά σε κάποιο dumping και δεν πρέπει νομίζουμε να εφαρμόζεται ο κανόνας των χαμηλότερων δασμών για τις πρώτες ύλε και τέλος είμαστε κατά της αρχής ότι που λέγεται shipping clause και που συζητήθηκε προηγουμένως γιατί μπορεί να απαιτηθούν περισσότερες αποστολές σε δύσκολους καιρούς, αλλά μπορεί και να μειωθούν περισσότερο τα κέρδη των επιχειρήσεων λόγω του ντάμπινγκ. Τέλος έχουμε ανησυχίες για την τάση που διαφαίνεται να μειωθούν οι πόροι που διατίθενται για την εμπορική άμυνα. Κατανοούμε ότι η κατανομή των πόρων είναι κάτι δύσκολο για όλους μας σε αυτήν την συγκυρία η βιομηχανία πρέπει να θεωρηθεί προτεραιότητα όμως. Και καταλήγω αγαπητέ μου πρόεδρε, στα πλαίσια της τωρινής κατάστασης και του αδιεξόδου στον ΠΟΕ, οποιαδήποτε μονομερής ε, ενωσιακή απόφαση μπορεί να στρεβλώσει την οικονομία. Μπορεί σε μια πρώτη φάση το κριτήριο, το ύψιστο κριτήριο να είναι η καλύτερη τιμή για το κάθε προϊόν, αλλά το μακροπρόθεσμο κριτήριο πρέπει να είναι η δίκαια τιμή για σταθερή ποιότητα. Πριν από μερικές, μετά από μερικές εβδομάδες θα κάνει την πρόταση της η Κομισιόν και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να το συζητήσουμε για να γνωρίζουν όλοι ότι είναι πολύ σημαντική για τη βιομηχανία, που σημαντικά για τη βιομηχανία αυτά τα εργαλεία εμπορική άμυνα. Ευχαριστούμε τώρα τα συνδικάτα, διότι και τα συνδικάτα είναι ενδιαφερόμενοι εδώ. Πολλές φορές μάλιστα είναι οι πρώτοι στόχοι και θύματα των αθέμητων παρακουτικών από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες. Ας τα ακούσουμε λοιπόν και αυτά. Έχουμε τον Θωμά Τζένκινς που είναι σύμβουλος στον γενικό, προς τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής ΓΕΣΕ. Έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν συμφορούμε σε μεγάλο βαθμό με τους κοινωνικούς μας εταίρους. Θέλω να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, για την συνέπεια μεταξύ βιομηχανικής πολιτικής και εμπορικής πολιτικής και δασμολογικής πολιτικής αφετέρου. Δεν είναι δυνατόν να δούμε το, τα, εμπορικά, τα μέσα εμπορικής άμυνας χωρίς να δούμε πώς εξελίσσεται η βιομηχανική περιοχή, ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολλοί λένε ότι ε, η Ευρώπη είναι το παγκόσμιο χωριό του τρελού, ε, ο παγκόσμιος ε, τρελός του χωριού, συγγνώμη. Ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, δεν μιλάμε για προτάσει ταυτικισμού, μιλάμε για ίδιε συνθήκε για όλου. Δεύτερον, οι ε, συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουν πολλά, υπάρχουν πολλά προϊόντα, άπειρα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται στην Κίνα ή από την Κίνα αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτά αυτό θα γίνεται χωρίς dumping και με ε, καλές κοινωνικές και εργατικές συνθήκες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, που αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας ότι ε, τα συνδικάτα έχουν, πολλά, έχουν μεγάλο διακύβευμα, έχουμε υποβάλει προτάσεις. Ο κ. Χοφμάιστερ ε, είπε ότι η ε, Κομισιόν δεν σκοπεύει να ακολουθήσει ορισμένα μέσα από τις ε, ιδέες μας, όμως μην ξεχνάτε ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε ένα μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το γεγονό ότι εμεί υποβάλαμε μία απάντηση ενώ τα λόμπι 300 δεν σημαίνει ότι η δική μα είναι μικρότερη αξία. Επίση, η δυνατότητα τα συνδικάτα να κάνουν καταγγελίες σε τέτοιους περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι, οι οποίοι δημοσίευσαν την έκθεσή τους τον περασμένο Φλεβάρι, ε, ήταν σαφεί. Ε, συμβούλευαν και σύστηναν τα συνδικάτα να έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελίες οι οποίε ενδεχομένω θα μπορούσαν να ερευνώνται αυτεπάγγελτα από την Κομισιόν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει κάτι τέτοιο. Ήδη γίνεται. Στην Αυστραλία και στι ΗΠΑ ε, τα συνδικάτα μπορούν να κάνουν καταγγελίε ε, κατευθείαν. Στη Νέα Ζηλανδία και την Νότια Αφρική τα συνδικάτα μαζί με του εργοδότε μπορούν να ξεκινήσουν να υποβάλλουν τέτοιε καταγγελίε. Βέβαια, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για μα ε, το πρώτο μοντέλο, αλλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ακολουθήσουμε ένα σύστημα ε, σύμφωνα με το οποίο μέσω των Επιτροπών Κοινωνικού Διαλόγου ή με κάποιο άλλο τρόπο θα συνεργαζόμασταν με την εργοδοσία για την υποβολή καταγγελιών. Ε, εμάς ε, δεν μας νοιάζει να μας, υποβάλουν, να μας επιβάλλουν αντίπεινα οι Κινέζοι, έτσι κι αλλιώς υποβάλλουν ακόμα και χωρίς να έχουμε υποβάλει εμείς καταγγελίες. Ε, Οπότε, αν η, αλλά, αν η εργοδοσία σε, συμμετείχε στην όλη διαδικασία, θα ήταν ακόμα πιο ισχυρές αυτές οι καταγγελίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ωραία. Ας ξεκινήσουμε την συζήτηση με τους άλλους παρόντες. Με, ξεκινώ με τη δική μου επιτροπή. Αν μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω αν έχουμε ίσες συνθήκες για όλους, η ίση μεταχείριση. Αλλά προτιμώ την επιτροπή μου καταρχήν. Ε... Φρανσίσκα Κέλλερ καταρχήν. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους παρουσιάζουν την άποψή τους. Ε, θέλω να θέσω δύο θέματα. Ε, για τη διαφάνεια, όλοι είμαστε υπέρ της διαφάνειας προφανώς, αλλά ε, μπορεί να γίνει ε, να στραφεί εναντίον μας. Στραφεί μάλλον εναντίον με την έννοια του ότι μπορεί να είναι υπέρ των συμφερόντων εξαγωγών που δεν έχουν σχέση με αυτούς που πλήττονται από το dumping. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, ε, θα θέλαμε να μικρύνει η προθεσμία για τα προσωρινά μέτρα, γιατί 9 μήνες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλά μπορούν να συμβούν, το είδαμε αυτό ε, με την, στην υπόθεση Κίνας PV. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πρόβλημα με την μικρή, το να μικρύνουμε την προθεσμία. Ο κανόνας του μικρότερου δασμού δεν ξέρουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε εμεί αυτή την πρακτική αν δεν μας ακολουθούν και οι υπόλοιπε χώρες. Και γιατί θα έπρεπε να εφαρμόζουμε αυτό τον ε, κανόνα σε χώρες οι οποίες ε, ακολουθούν πρότυπα χαμηλότερα από τα δικά μας, χαμηλότερα από το ελάχιστο. Ε, επίσης, ε, ε, δεν ε, θέλουμε να, μάλλον να συμπεριληφθούν και οι θηγατρικές ε, εταιρείες εταιριών που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα, στα οποία δεν αναφέρεται η πρόταση της Κομισιόν ιδιαίτερα για παράδειγμα, οι πιο εύκολε ε, διαδικασίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα το υποστηρίζαμε γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δυσκολεύονται πολύ αυτή τη στιγμή, που υποβάλουν καταγγελίες. Δεύτερον, το, το κοινωνικό και περιβαλλοντικό dumping. Πρέπει να ορίσουμε την βλάβη με πιο ευρύ τρόπο, έτσι ώστε να αναγνωριστεί του να γνωριστεί η παρουσία και μεγαλύτερων προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή. Τέτοιου είδους ε, παγκόσμια προβλήματα έχουν ε, οικονομικό υπόβαθρο και οι ζημίες που προκύπτουν, οι βλάβες που προκύπτουν ε, είναι πολύ συχνά ε, λιγότερο απτές. πολύ συχνά ή ε, το περιβαλλοντικό dumping ισοδυναμεί με επιδότηση. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να τα δούμε στο πλαίσιο του ότι και οι κανόνες για τις επιδοτήσεις θα πρέπει να ρυθμιστούν σε επίπεδο ΠΟΕ. Ε, τώρα, ε, σε ό,τι αφορά την ηλική, τον ορισμό της ηλική βλάβης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μη συμμόρφωση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, ε, καθώς και ε, επίσης η χρηματοδότηση για την επιτυχία ε, περιβαλλοντικών στόχων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει οθεί στην Κομισιόν να ηγηθεί του υπόλοιπου κόσμου στον ΠΟΕ, έτσι ώστε να, ληφθεί υπόψη, να ληφθεί υπόψη η συνέπεια τη κλιματική αλλαγή και να εξυγχρονιστεί το σύστημα. Γιατί αν θέλουμε ε, πραγματικά να εξυγχρονίσουμε ε, τους κανόνες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις καινούριες προκλήσεις που εμφανίζονται. Ε, υποστηρίζουμε την πρόταση τα συνδικάτα να μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες επίσης να συμμετάσχουν στενά στην ακριβή αξιολόγηση της βλάβης για παράδειγμα που έχει πάρει τη μορφή απολύσεων. Τέλος, ε, απογοητεύομαι που η Κομισιόν προτείνει παράταση της ε, προθεσμίας για τις ε, ε και για την επιβολή ε, μέτρων Ε, θα, το θέμα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του πακέτου Omnibus. Ε, ευχαριστώ πολύ. Περιμένω την απαντήσει. Ο πρόεδρος. Κυρία Κιαλέ, πάντοτε είμαι πρόθυμος να σας δώσω περισσότερο χρόνο. Γιατί όποια και να είναι, να είναι οι διαφωνίες μου, πάντοτε οι διαφωνίες μας Πάντοτε θαυμάζουμε τη δέσμευσή σας, την προετοιμασία σας και τη σοβαρότητα με την οποία συμμετέχετε στις εργασίες μας. Αλλά την επόμενη φορά θα σας περιορίσω το χρόνο. Έχω 7 ομιλητές από τη δική μου επιτροπή και πρέπει να αφήσω και χρόνο στο ακροατήριο. Δύο λεπτά λοιπόν και το πρώτο θύμα είναι ο Helmut Scholz. Πρέπει λοιπόν να είμαι σύντομος πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι συμφωνώ αρκετά με αυτά που είπε η κυρία Κέλλερ αλλά ομολογώ ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τη γενική αυτή προσέγγιση. Γιατί βλέπω εδώ στην αφίσα μία ασπίδα. Δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που έχουμε θέσει. Είμαστε εκτός θέματος. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία απαιτεί νέες απαντήσεις, όχι οι απαντήσεις του παρελθόντος, τα θέμα των πρώτων υλών. Τι χρειάζεται δηλαδή για την παραγωγή μας. Και άρα η απάντηση πρέπει να είναι ότι και οι εμπορικοαμυντικοί μηχανισμοί πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόκληση. Γι' αυτό απαντώ ότι πράγματι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό dumping και τις επιχορηγήσεις που πρέπει να έχουν ορισμένες χώρες για τον ανταγωνισμό τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσω ότι και αυτό αφορά και τα συνδικάτα που κατανοώ τα αιτήματά τους, ό,τι λέγω ότι πρέπει να απαντήσουμε, να ανταποκριθούμε και στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, αυτό το εργαλείο εμπορικής άμυνας πρέπει να το αντιμετωπίζει και αυτό. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν, ρε, ρωτώ την Κομισιόν, θεωρείται ορισμένα κριτήρια από αυτά που ανέφερα ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στην πρότασή σας. Τέλος, τα μέσα που έχουμε, που πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτό το εργαλείο πρέπει να αναφέρουν και το πώς, με ποιο τρόπο θα δούμε το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας στην βιομηχανική ανάπτυξη. Παράδειγμα, για την ηλιακή ενέργεια και τις πρωτοβουλίες της Κίνας επ' αυτής. Γιατί εδώ έχουμε χάσει. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι το εργαλείο αυτό στην πρόταση της Κομισιόν πρέπει να ενσυγχρονιστεί προς τον 21ο αιώνα. Ξεπεράστε το χρόνο σας. Τώρα η κυρία Μπέλα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ε, προλαλήσαντες. Θέλω να τοποθετήσω το θέμα στην σημερινή συγκυρία. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης Μιλάμε για μια Ευρώπη που ζει μια μαζική αποβιομηχάνηση. Οπότε είναι σημαντικό να τοποθετήσουμε όλο το θέμα αυτό στη σημερινή συγκυρία. Γιατί άλλη κατάσταση σήμερα, άλλη όταν η Κομισιόν ξεκίνησε τη διαβούλευσή της. Ε, μιλάμε για εξυγχρονισμό, μιλάμε για αναθεώρηση του κανονισμού Όμω κατά τη διάρκεια τη διαβούλευση, ε, διαφάνει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύει πως το σύστημα είναι αποτελεσματικό διότι μόνο το 25% απάντησαν ότι είναι μη αποτελεσματικό. Σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό, ε, δεύτερο σχόλιο μου, δεν θα πρέπει ο εξυγχρονισμό να ιδωθεί ως ε, χαλάρωση των διαθέσιμων μέσων γιατί κάτι θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη κατάρρευση ε, ή μη εφαρμογή των μέσων τη στιγμή που ε, χρειαζόμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία. Για παράδειγμα σκέφτομαι ιδιαίτερα στην Κίνα. Ε, θα πρέπει να πιστεί να ασκεί ένα πιο θεμητό εμπόριο. Δεν θα πρέπει η αναθεώρηση να αποτελεί αποδυνάμωσή μας. Σε ό,τι αφορά την χρήση των μέσων αυτών, η χρήση θα πρέπει να είναι δίκαιη, ε, αιτιολογημένη, θεμητή και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αναζητηθεί ένας τρόπος να είναι εύκολη η εφαρμογή των μέτρων, μέσων. Και υπό αυτό το πνεύμα έγινε και η διαβούλευση. Όταν είναι δικαιολογημένη, αιτιολογημένη η ε, χρήση αυτών των μέσων, θα πρέπει η Κομισιόν ε, να μπορεί να αντιδράσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο, με τεχνικά και οικονομικά μέσα. τρίτον, ε, για τις αυτεπάγγελτες διαδικασίες ε, που έχουν τη θέση τους, έχουν δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, αποφεύγουμε μια βαριά και περίπλοκη διαδικασία ε, καταγγελίας και δεύτερον, αποφεύγουμε τα αντίπεινα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για τη διαφάνεια. Θέλω μόνο να θέσω το ερώτημα της αναθεώρησης αυτού του κανονισμού γιατί δεν ε, τον ενημερώσαμε, δεν τον επικαιροποίησαμε απλώς. Από το 1995 έξι φορές έχει γίνει επικαιροποίηση του κανονισμού, όχι η πλήρης αναθεώρησή του όμως. Μπορείτε επίσης να μας εξηγήσετε γιατί τα μέτρα ε, αυτά τα οποία προτείνονται θα μας εγγυηθούν καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των μέσων. Τελευταία ερώτηση, ε, ποιο είναι το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να διατηρεί τον κανόνα του ε, μικρότερου δασμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους τους προλαλήσαντες. Ε, τρεις παρατηρήσεις καταρχήν η ε, προθεσμία ανάμεσα στην κατάθεση της ε, ε, και την λήψη των μέτρων είναι πέντε φορέ ε, μεγαλύτερες, πέντε φορές μεγαλύτερη από τις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη πρέπει να μείνουμε 9 ως 12 μήνες για τους δασμούς, για την επιβολή δασμών οι ίδιοι δασμοί είναι 35% στην Ευρώπη κατά μέσο όλο, 130% στις ΗΠΑ, τέσσερις φορές λιγότερο. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφαρμόζει τη διαδικασία, την αυτοπάγγελτη δηλαδή διαδικασία. Ε, αυτή την έννοια δεν θα με πειραζε ένας εξυγχρονισμός των μέσων, αλλά όχι για να τα αποδυναμώσουμε αυτά τα μέτρα. Ε, θα Νομίζω ότι 80% των βιομηχανών μας ε, συμφωνούν με αυτό. Ε, δεν ε, θα πρέπει να υποχωρήσουμε εναντί των σειρών του προστατευτισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει όμως ένα επαρκές οπλοστάσιο που θα μας επιτρέπει να έχουμε περιθώριο δράσης και θα μας βοηθήσει να καταστήσουμε τις παγκόσμιες οικονομικές αλλαγέ πιο θεμητές. Ε, δεν θα πρέπει να ε, επιτρέψουμε ε, σε κάποιες χώρες να έχουν πρόσβαση στις αγορές μας με χαμηλά πρότυπα εργασιακά, τιμωρικά κλπ. Ε, έχουμε, θα έχουμε μέλλον στην Ευρώπη μόνο αν μπορούμε να υπερασπίσουμε ε, την βιομηχανία μας από θέμητες πρακτικές, για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά. 15% ε, των ερευνών γίνονται, αφορούν θέματα επιδοτήσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίση διαπιστώνω ότι οι Πολιτείε ε, έχουν δύο φορέ μεγαλύτερο προσωπικό που χρησιμοποιείται για θέματα αντιεπιδοτήσεων και εναντίον του dumping. Αυτό βοηθάει πολύ περισσότερο βέβαια. Ε, αν ε, η χρήση περισσότερου προσωπικού και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας επέτρεπε να γλιτώσουμε μερικά εκατομμύρια στη βιομηχανία, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το προσωπικό. Τέλος, ε, τα μέσα που διαθέτουμε δεν είναι, λίγο αδύναμα. Αλλά, ε, εν πάση περιπτώσει, ε, ποια είναι τα συμπεράσματα που έβγαλε η Κομισιόν από την προσπάθεια μεταρρύθμισης του 2006, πώς μπορούμε να προσανατολίσουμε, προς τα πού θα προσανατολιστεί η πρόταση Κομισιόν και τέλος, ε, θεωρείτε ότι τα μέτρα αντιεπιδοτήσεων θα είναι πιο προσβάσιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος πάλι από το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή, όμως θα ήθελα να τονίσω ότι εκπλήσωμε που παρουσιάζεται αυτή η νέα προσέγγιση του συγχρονισμού των ε, μέσων άμυνας του εμπορίου ε, και πιστεύω ότι αυτό αντιφάσκει στις ε, παρελθούσες δηλώσεις του Επιτρόπου κ. Ντεγκούχτ. Και τώρα θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα. Ε, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε ε, μια μεγάλη οικονομική κρίση και επειδή υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης αυτών των αυτού του μηχανισμού, η Κομισιόν θα πρέπει να προβλέπει μέτρα τα οποία θα αναζωογονήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία, θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Και τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι ισόρροπα και θα πρέπει εν τέλει να καταλήξουν στην αποδυνάμωση των μέσων εμπορικής άμυνας προς ε, όφελος ε, των ε, εισαγωγέων-εξαγωγέων. Όσον αφορά τη διαφάνεια τώρα, η Κομισιόν προτείνει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται η προσωρινή δασμολόγηση εγκαίρως όμως ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να οδηγήσει στην ε, παράκαμψη αυτών των μέτρων ε, με το να δημιουργούν μεγαλύτερα αποθέματα οι εμπορευόμενοι. Τα αντίπεινα επίσης ε, και αντίμετρα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Είναι αντίπεινα τα οποία συνήθως προκύπτουν για πολιτικούς λόγους. Και η Κομισιόν προτείνει να αντιμετωπίσει αυτή την τάση με, την, με το να ξεκινάει ε, αυτεπαγγέλτος προσφυγές ε, που θα καταλήξουν ενδεχομένω σε επιβολή κυρώσεων. Είναι λοιπόν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα τα αντίμετρα από την Κομισιόν προς όφελό της. Όσον αφορά ε, της, την αναθεώρηση ε, δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί και σύγκριση με, ε, με προσφυγές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη όλα τα μπορούν να οδηγήσουν στη συντόμευση του χρόνου επεξεργασίας. Και επίσης όσον αφορά την επιβολή αυτού του μικρότερου δασμού ως ποινή, πιστεύω ότι θα οδηγήσει αρνητικά τελικά στην αύξηση δασμών που δεν είναι πάντοτε ένα χρήσιμο αποτέλεσμα αν επιβάλλονται ως κυρώσεις. Ε, και εν πάση περιπτώσει θα βοηθήσει τις χώρες που κάνουν μεγαλύτερες εισαγωγές και όχι τους τομείς και θα είναι και πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό. Ο πρόεδρος και τέλος ο Τζαν Λούκας. Ε, παρόλο ότι έχουμε λίγο χρόνο, ε, με βοηθάει το ότι ορισμένε από τι ερωτήσει μου έχουν ήδη γίνει από άλλου συναδέλφου. Θα περιστώ σε ορισμένε παρατηρήσει. Μία ένα από τα θέματα που προκύπτει πάντοτε είναι το εξής. Ε, θα πρέπει ε, να θα πρέπει οι προτάσεις μας να βασίζονται σε διαβούλευση διότι ε, ζούμε ένα μια παράξενη εποχή αντιφατική η κατάσταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας έρχεται σε αντίθεση μπορεί να μας οδηγήσει μάλλον σε προστατευτισμό ενώ η πολιτική μας γενικά είναι αντίον του προστατευτισμού. Η... Παρ' όλα αυτά έχουμε τομείς της οικονομίας μας που προχωράνε μπροστά και καινοτομούν. Θα πρέπει λοιπόν να Ε, λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το 80% των ερωτωμένων, ερωτουμένων ε, ανησυχούν. Ε, και στην προηγούμενη θητεία της ε, Κομισιόν ετέθησαν τα ίδια θέματα και η Κομισιόν είχε αποσύρει την πράσινη βίβλο ε, για τα μέσα εμπορικής άμυνας ε, διότι ήταν ε, πολύ υπερβολικά μάλλον νεοφιλελεύθερα. Συνεπώς πιστεύω ότι όταν περάσουμε από τη φάση διαβούλευση στη φάση της υποβολής προτάσεων ε, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τους, ερωτισμού, τους ε, ορισμούς, ε, την διαφάνεια, την ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων αντι-dumping, μεγαλύτερη επιλεκτικότητα και θα πρέπει όλα αυτά να τα εντάξουμε και στις εμπορικές μας συμφωνίες. Θα πρέπει επίσης ε, να καταπολεμήσουμε, να ε, αμυνθούμε μάλλον έναντι ε, των αντιπίνων που επιβάλλουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη σήμερα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που είχε υπόψη της η Κομισιόν όταν ξεκίνησε η διαβούλευση. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ενισχύ αυτή τη στιγμή. Ο φιλελευθερισμός, η απελευθέρωση φοβίζει και από την άλλη μεριά έχουμε την ανάγκη να καινοτομήσουμε. Υποτίθεται ότι θα τελειώναμε σε 40 λεπτά. 30 λεπτά λοιπόν για τους ομιλητές και 10 λεπτά για τις ερωτήσεις αλλά σύντομα Well, the gentleman from the Italian representation, yes, with a very short remark. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση από την Ιταλική Αντιπροσωπεία. Όχι πάνω από ένα μισή λεπτό, παρακαλώ. Thank you. It is really necessary to modernize... Είναι σημαντικό να εξυγχρονιστούν τα μέσα εμπορική άμυνα αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εγώ χαίρομαι για τη δημοκρατική προσέγγιση που υιοθέτησε η Κομισιόν αυτή τη φορά που προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο το θέμα αυτή τη φορά. Ε, όχι όπως ο κύριος Μάντελσον το 2006. Η Ιταλία τότε είχε μπλοκάρει τις προτάσεις, ευτυχώς. Ε, τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης είναι σαφή όμως. Πρώτον, η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών ε, είναι ε, δεν είναι εισαγωγή εξαγωγή, αλλά βιομηχανή. Δεύτερον, η πλειοψηφία είναι υπέρ τη ενίσχυση τη νομοθεσία για να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τρίτον, ε, τα TDI δεν είναι μέσα προστατευτισμού. Είναι το μοναδικό μέσο που έχουμε για την καταπολέμηση του αθέμη του ανταγωνισμού. Η ισχυρότερη νομοθεσία για τα μέσα αυτά σημαίνει μεγαλύτερη ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορική της πολιτική και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, στον ΠΟΕ βρισκόμαστε σε κρίση, το γνωρίζετε. Συνεπώς αυτό που προτείνουμε είναι ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική νομοθεσία ε, μέσων εμπορικής άμυνας χωρίς ε, το τεστ της, ε, των συμφερόντων της κοινότητας, χωρίς τον κανόνα του, μειωμένου, του ε, μικρότερου δασμού. Όπως οι ΗΠΑ, όταν υπάρχουν αθέμητες πρακτικές θα πρέπει τα μέτρα να εφαρμόζονται αυτόματα. Ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από ένα τέτοιο αυτόματο σύστημα τα μέσα εμπορική άμυνα είναι τεχνικά μέσα. Δεν θα πρέπει να πολιτικοποιηθούν. Αν είχαμε αποτελεσματική νομοθεσία που να υποστηρίζει τη βιομηχανία μα, όπω προτείνουμε, θα μπορούσαμε να δώσουμε και καθεστώ οικονομία αγορά αυτόματα στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει νομική διατάξη που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλο μέλο του ΠΟΕ ε, ε, μέχρι το 2016. Η ζητούμε από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή επαναβιομηχάνηση ε, μέσω της ενίσχυσης όμως των μέσων εμπορικής άμυνας. Θα πρέπει να αποφύγουμε επίσης τα κόλπα της Κομισιόν. Παρακαλώ τελειώνετε λέει ο Πρόεδρος και χρειάζομαι και το όνομά σας για τα πρακτικά. Αμαντέο τέτη από την Ιταλική κυβέρνηση. Περνάμε στην Eurocommerce. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, αντιπροσωπεύει 6 εκατομμύρια ε, εταιριών χονδρικής και λιανικής. Ε, δεν νομίζω ότι μας εκπροσώπησε η Business Europe, οπότε θέλω να κάνω μερικές δικές μας παρατηρήσεις. Το σημαντικό είναι να μην επαναλάβουμε το σενάριο του 2007 με σύγκρουση ανάμεσα στα συμφέροντα της ε, βιομηχανίας και ε, τα, στα συμφέροντα των εισαγωγέων. Πρέπει να βρούμε μια λύση που επικοδομητικά θα ξανασυμφιλιώσει ε, τις διαφορετικές θέσεις εισαγωγέων και βιομηχάνων ε, κατασκευαστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα από ό,τι πριν από πέντε χρόνια μέσω του διαλόγου. Ε, το βασικό σημείο για μας είναι, δεδομένου ότι το αντι είναι ε, προς ε, και των εισαγωγείων και των ε, βιομηχάνων ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ρήτρα αποστολής. Επίσης, κατευθύνσεις γραμμές για τη δοκιμή του, των συμφερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι ε, αυτεπάγγελτες έρευνε δεν είναι καλή ιδέα και ο κανόνας του μικρότερου δασμού είχε νόημα στο παρελθόν και πιθανότητα θα έχει, μέλλον, ε, θα έχει νόημα και στο μέλλον. Ε, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ακρόαση ή κατάθεση απόψεων. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Ρενέ Φαν Σλότεν. Αντιπροσωπεύω την χημική βιομηχανία της Ευρώπης. Η βιομηχανία μας θεωρεί ότι το παρόν σύστημα είναι πολύ ισορροπημένο. Είμαστε μια βιομηχανία που εξάγει παραπάνω από ε, χημικά αξίας άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ και εισάγουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, εμπορεύματα αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ ισορροπημένοι σε ό,τι αφορά το dumping. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα ε, με προστατευτικό τρόπο. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι ότι υφίσταται μια στρέβλωση ε, εξαιτίας των εξαγωγικών δασμών, εξαγωγικών περιορισμών, διπλών τιμών για τις ε, κλπ. Αυτές, αυτές οι στρεβλώσεις ε, δεν αντιμετωπίζονται ε, σωστά μέσω των συμφωνιών ελευθερομπορίου ούτε από τον ΠΟΕ. Ούτε, ούτε καν με τον, κανονισμό, τον νέο κανονισμό για τις, το τις προτιμήσεις, τον κανονισμό. οπότε, τον κανονισμο την dumping δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ε, διατάξεις, μάλλον θα πρέπει να συμπεριλάβουμε διατάξεις που να καθιστούν σαφές ότι όταν υπάρχουν στρεβλώσεις ε, σε σχέση με τις πρώτες ύλες θα λαμβάνονται μέτρα. Ε, τέλος, ε, πολλοί αναφέρθηκαν στο κοινωνικό και το περιβαλλοντικό dumping. διαφωνώ ρητά και κάθετα με την προσπάθεια να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο στα ε, μέσα εμπορικής άμυνας. Χρειαζόμαστε ε, ένα κανονισμό ισορροπημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να προσπαθήσουμε ε, να ε, επιβάλλουμε κοινωνικές ε, πρακτικές μέσω διορθωτικών μέτρων στα σύνορα. Με, μέσα δηλαδή που έχουν σχέση με την, το εμπόριο εκπομπών κλπ. Ευχαριστώ. Also put... Άλλος κανείς? Ε, ήρθε η σειρά μου. Έχω και εγώ τώρα τι ερωτήσεις μου την Κομισιόν. Αναφέρθηκε η προσέγγιση του Επιτρόπου κ. Ντεγκούχτ και αναρωτιέμαι γιατί η Κομισιόν αποφάσισε να ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία. Δεύτερον, στο κείμενο της Κομισιόν αναφέρεται ότι ο, σκοπό, ο στόχος είναι να αυξήσει την ευελιξία, επιλεξιμότητα και δεν φοβόσαστε ότι μπορεί να κατηγορηθείτε, να κατηγορηθείτε ότι έχετε μια κρυφή ημερήσια διάταξη, μια κρυφή ατζέντα. Είναι κατάλληλη η στιγμή αυτή για την μεταρρύθμιση τώρα που βρισκόμαστε μέσα σε μια μεγάλη κρίση. Αντί δηλαδή να στείλουμε ένα μήνυμα περισσότερης ευελιξίας στα, μέσα, στα μέσα του εμπορίου. Προσπαθούμε τώρα να τα ενισχύσουμε περαιτέρω. Έχω εδώ μία ανακοίνωση τύπου της Αυστραλίας πριν από δύο εβδομάδες, 4 Δεκεμβρίου, και λέει «Ενίσχυση του συστήματος anti-dumping της Αυστραλίας». Και στα μέτρα περιλαμβάνονται η δημιουργία ενός συμβούλου που θα χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Προπολογισμό της Αυστραλίας για να βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις προσφυγές που γίνονται για αντι-dumping. Δεν πιστεύετε λοιπόν υπό τις παρούσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει κάτι εδώ που μας υποδεικνύει ότι τα TDIs θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντί να είναι τόσο δαπανηρά ώστε να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Διότι οι προσφυγές είναι τόσο χρονοβόρες και ακριβές. Και όσον αφορά τώρα τις εσωτερικές υπηρεσίες της Κομισιόν. Ποιες είναι ακριβώς ε, το διαθέσιμο δυναμικό Όσον αφορά τι υπηρεσίε τη Κομισιόν για την παρακολούθηση του anti-dumping, βρισκόμαστε, βρισκόσαστε στην Κομισιόν υπό τρομερή πίεση και δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις προσφυγές αυτές. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω τι ακριβώς κάνει η Αυστραλία πριν από δύο εβδομάδες. Αποφάσισαν να διαθέσουν πολύ περισσότερους πόρους και εμπειρογνώμονες που θα χρηματοδοτηθούν για την πολιτική αντι-dumping. Και επιπροσθέτως Εκτός από αυτά που αποφάσισαν να διαθέσουν, 24,4 εκατομμύρια θα διαθέσουν για αυτή την πολιτική μέχρι το 2016 για να εξασφαλίσουν ότι το σύστημα αυτό μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσει της ε, οικονομίας και βιομηχανίας της Αυστραλίας και για να μπορέσει να ξεπεράσει τις μεγάλες καθυστερήσεις που δημιουργούνται μέσα σε αυτό το σύστημα καταπολέμησης αντι-dumping με τον όγκο των κανονισμών. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι αντί να λανσάρετε και να ξεκινήσετε μία μεταρρύθμιση του μηχανισμού θα πρέπει να τον καταστήσετε πιο ευέλικτο και πιο εύχριστο. Αυτή είναι η ερώτηση στην οποία θα ήθελα πολύ η Κομισιόν να απαντήσει. Και τώρα δίνω το λόγο με αντίθετη σειρά στους ε, ομιλητές του, του πάνελ μας. Thank you very much, Mr. Chairman. I am uh, going to be very brief. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. In the first place, I think we must make a Θα είμαι σύντομος. <laughs> Ε, θα πρέπει καταρχάς να κάνουμε διαχωρισμό σε αυτή τη συζήτηση μεταξύ του να παίζουμε με τους υπάρχοντες κανονισμούς και τη δημιουργία νέων κανονισμών που θα μας θέσουν σε πορεία σύγκρουσης με τις υποχρεώσεις μας των ΠΟΕ ως έχουν. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό και φρόνιμο να δούμε την άσκηση αυτή, αυτή σαν ένα είδος προληπτικό χτύπημα πριν, ε, κάνουμε τις, ε, πριν αρχίσουν οι διαβουλεύσεις στη Γενέβη. Δεύτερον, Έχουμε στην ε, πρόταση, αν μου επιτρέπετε να πω πρόταση της Κομισιόν, ε, μία σειρά ευέλικτων στοιχείων που προτείνονται, αλλά οι ευέλιξίες αυτές είναι ε, μονομερείς θα έλεγα. Υπάρχουν ευελιξίες και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Και όπως λέτε, αυτή η ρήτρα μεταφορά στο shipping clause, τη βρίσκω πολύ περίεργη πρόταση, πρέπει να ομολογήσω. Αυτή η καημένη εισαγωγή και εξαγωγή θα αντιμετωπίσουν, με, θα αντιμετωπίσουν προσωρινούς δασμούς τελείως αναπάντεχους, ουρανοκατέβατους, όπως λέμε, όταν μία απόφαση ε, μεταφοράς από έναν εξαγωγέα προϊόντων έχει ληφθεί πριν από 9 μήνες και θα πει ότι πού να φανταστώ εγώ ότι τελικά θα επιβληθούν ε, δασμοί αντι-dumping. Ε, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ψευδές τεχνητό μέτρο. Και εκεί που επιμένω ιδιαίτερα είναι ότι βεβαίως έχουμε νέες προκλήσεις που δεν υπήρχαν παλιότερα όμως, το ερώτημα είναι εάν οι κανόνες ως έχουν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Και εγώ δεν άκουσα κανένα επιχείρημα μέχρι τώρα για την αλυσίδα προμηθειών που είναι ένα επιχείρημα το οποίο προβάλλεται σε αρκετά έγγραφα. Υπάρχει όντως ανάγκη να αλλάξουν οι κανόνες για να αντιμετωπίσουμε, για να χειριστούμε, εν πάση περιπτώσει, την αλυσίδα προμηθειών. Δεν υπάρχει ανάγκη. Διότι το θέμα αυτό μπορεί να το καλύψουν σαφώς οι, οι, οι σημερινοί κανόνες. Το ερώτημα είναι σαφές. Ποια είναι η προέλευση του προϊόντος και καλύπτεται αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο Δόκτωρ Βέρμουλς. Ευχαριστώ. Μερικά σύντομα σχόλια. Καταρχάς, μετά από αυτά που είπε ο συνάδελφός μου εκ δεξιών, συμφωνώ απολύτως ότι από διεθνή άποψη μπορεί κανείς να υιοθετήσει τους κανόνες που ΕΣΥΝ, WTO+, δεν μπορεί κανείς να πάει λιγότερο από τον ΠΟΕ. Δεν μπορεί κανείς να εφαρμόσει κανόνες χαμηλότερους από τον ΠΟΕ. Που σημαίνει ότι είτε το θέλουμε είτε το, ή δεν το θέλουμε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα TDIs εναντίον του κοινωνικού dumping, εναντίον του περιβαλλοντικού dumping. Εάν θέλουμε να πολεμήσουμε αυτού του είδους το dumping, τότε πρέπει να βρούμε μηχανισμούς άλλους, αλλά όχι στον τομέα των μέσων εμπορικής άμυνας. Γιατί έτσι ακριβώς συμμορφωνόμαστε με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει με τον ΠΟΕ. Τρίτον, όπου ο εκπρόσωπος της ETAC, ETUC δηλαδή, είπε ότι μπορούμε ίσως να χειριστούμε τα θέματα αυτά με διεθνούς κανόνες και όχι με τους κανόνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ευρωπαϊκή Νομολογία. Εάν λοιπόν μπορούν να υιοθετηθούν οι διεθνείς κανόνες, οι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καλώς να χρησιμοποιηθούν. Εάν έχουμε κοινωνικό ή dumping. Τέταρτον, και πρώτο τελευταίο, ε, όσον αφορά την διπλή τιμολόγηση και εξαγωγική δασμή που ανέφερε ο κύριος Φεσλόιτεν, Υπάρχουν ήδη μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα και η Κομισιόν στο πλαίσιο του αντι-dumping μπορεί επαρκώς να αντιδράσει όταν ε, βρει έναν μηχανισμό διπλής τιμολόγησης ή dumping, ε, διότι τα αποτελέσματα θα ήταν χειρότερα αν αρχίσουμε να λειτουργούμε υπό ένα διαφορετικό σύστημα. Όταν λοιπόν επισημανθεί μια τέτοια κακή πρακτική, μπορεί η Κομισιόν οπωσδήποτε να δράσει μέσα στο πλαίσιο των TDIs. Και εδώ, σε αυτό το τελευταίο μου σημείο, διαφωνώ με τον Ζακ Μπουρζουά όσον αφορά την αλυσίδα προμηθειών. Υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι έχουμε δει περιπτώσεις ήδη στο παρελθόν και θα δούμε και άλλες στο μέλλον, όπου παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη πλευρά παραγωγή στην Κίνα ή στην Κορέα κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, κατά 90% δηλαδή Δηλαδή κάνουν την παραγωγή σύμφωνα με τους μετρήσιμους όρους ε, προέλευσης και καταγωγής χώρας και υπήρχε ακριβώς αυτή η υπόθεση για τη συναρμολόγηση των μόντεμ στην Κίνα. Δεν μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει, να παραπέμψει κανείς σε κανόνες προέλευσης για να κατηγορήσει την Κίνα. Ε, οι κανόνες προέλευσης δεν καλύπτουν αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συζητούμε μια πρωτοβουλία της Κομισιόν, επομένως σωστό είναι ο τελευταίος λόγος να ανήκει σε εκείνη. Ευχαριστώ καθηγητά Μορέρα και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και τα για τα ενδιαφέροντα πράγματα που είπαν. πολλά ερωτήματα αφορούσαν ακριβώς τη ρίζα του προβλήματος, τους στόχους μας δηλαδή. Θα ήθελα να απαντήσω σε μερικούς από τους βουλευτές και σε εσάς τον ίδιο. Όπως είπε και ο Ιταλός εκπρόσωπος δικαίως, έγινε προσπάθεια πριν από πέντε χρόνια από τον Επίτροπο Μάντελσον που δημιούργησε μεγάλες αντιθέσεις Τόσο πολλές που τελικά δεν τη συνέχισε. Αντίθεση μεταξύ δύο ομάδων χωρών το Ηνωμένο Βασίλειο ήθελε να συνεχιστεί η προσπάθεια, άλλες όχι. Αλλά υπήρξε τόσο μεγάλη διαφορά στο Συμβούλιο που σταμάτησε η προσπάθεια και αυτή η αντίφαση αντικατοπτρίστηκε και σε κόλπους της βιομηχανίας. Τώρα, τι συμπεράσματα να βγάλουμε από αυτό. Ο Επίτροπος Ντοχούχτ έχει δεσμευτεί να εξυγχρονίσει με διατήρηση της ισορροπίας. Γι' αυτό διατύπωσε τα πράγματα έτσι όχι απλώς ενδυνάμωση γιατί αυτό θα ερμηνευθεί αρνητικά. Εμείς θέλουμε να διατηρηθεί η ισορροπία. Να υπάρξει μια εξισορρόπηση δηλαδή μεταξύ των συμφερόντων των εισαγωγέων και της βιομηχανίας. Αυτά προσπαθεί να κάνει η Κομισιόν και αντιμετωπίζουμε τώρα πιέσεις πολιτικές από τρίτες χώρες, αλλά ο Επίτροπος Δεχούχτ προσπάθησε να εφαρμόσει το δίκαιο, το ισχύον δίκαιο. Αυτό το δρόμο θέλει να ακολουθήσει. Έτσι, θέματα όπως η διαφάνεια, η προβλεψιμότητα και η εμπιστοσύνη όλων των χριστών διασφαλίζονται. Αυτό σημαίνει ένομη διοίκηση. Αυτό θέλω να το πω πολύ ρητά. Τώρα, πώς θα το πετύχουμε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν μερικά τεχνικά προβλήματα που δεν μπορώ να τα θίξω όλα. Μερικά όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διαφάνεια. Συζητήσαμε ήδη το ότι η πληροφόρηση δεν αποδυναμώνει το μηχανισμό δίνει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να αντιδράσουν. Και δεν είναι αποδυνάμωση αυτό. Θα μπορούσε κανείς να συζητήσει θέματα περιόδων και κλπ. Αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Τα αντίμετρα είναι άλλο πραγματικό θέμα και αυτά που προτείνουμε απαντούν σε κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Τώρα η δράση. Έχουν ακουστεί εδώ δύο απόψεις. Η Business Europe είπε ότι ο κανόνας για τη μείωση των δασμών θα χρειάζεται περισσότερες εξαιρέσεις. Ενώ άλλοι και μεταξύ των εμπειρογνωμόνων λένε όχι τα πάτε πολύ μακριά τα πράγματα να μην πλήξετε τις τρίτες κυβερνήσεις αλλά τις εταιρείες εμείς θέλουμε να υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις αλλά όχι γενίκευσή τους. Για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα άκουσα ότι ο καθηγητής Μπουρζουά θεωρεί ότι είναι θέμα κατεξουσιοδότηση πράξεων που πρέπει καλύτερα να τις καθορίσει ο νομοθέτης. Μπορεί ο νομοθέτης να ζητήσει καλύτερο ορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, αλλά σε εμά πάλι θα μεταφέρει η δικαιοδοσία για την εφαρμογή. Εγώ με μεγάλη χαρά άκουσα ότι όλοι θέλουν να υπάρξει καθορισμός κατευθυντηρίων γραμμών και αυτό ακριβώς κάνουμε. Για το πολύ σημαντικό θέμα των συνδικάτων τώρα. Think currently, uh, when the... Αν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός από κοινού Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε τα συμφέροντα των συνδικάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί, φανταζόμαστε, τα συμφέροντα της ε, κάποιας εταιρείας. Αλλά αν υπάρχει κάποιο παράπονο το οποίο στηρίζουν μόνο τα συνδικάτα και όχι και το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί κανείς να υποψιαστεί ότι πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα. Αν όμως βρεθεί κάποιο σύστημα διαφορετικό, τότε ο Επίτροπος είναι ανοιχτός σε άλλες ιδέες, ίσως για τις κοινέ υποβολές παραπώνων. Για τον ορισμό της επιχορήγησης, η κυρία Κέλλερ μας είπε τι είναι επιχορήγηση ή πότε χρειάζεται επιχορήγηση, ας πούμε, αν κανείς δεν αντιδράσει για την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών. αυτά δεν τα λέει ο ΠΟΕ. Η επιχορήγηση είναι ένα χρηματικό ποσό που χορηγείται για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο καθηγητής Μορέιρα, ε, καθηγητά Μορέιρα είμαστε στο πλευρό σας. Υπάρχει ήδη το Help Desk των μικρομεσαίων και αυτό μπορούμε να το επανεξετάσουμε. Δεν θέλουμε να αποκλειστούν οι μικρομεσαίες από τη χρήση του μηχανισμού. Και τώρα οι πόροι, αν ζητήσετε περισσότερους πόρους για τη γενική μας διεύθυνση, φυσικά θα είμαστε υπέρ, αλλά πέστε το στα κράτη-μέλη που μιλούν για 5% μείωση των λειτουργικών εξόδων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Μου άρεσε πολύ αυτό το εργαστήριο. Νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση και τέθηκαν όλα τα προβλήματα. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω τα βασικά. Πρώτον, ο μηχανισμός εμπορικής άμυνας δεν είναι αποκλειστική δικαιοδοσία της Ένωσης. Οι συνθήκες μιλούν για ελεύθερο και θεμητό ανταγωνισμό, δίκαιο. Και επομένως έμεσα υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Δεύτερον, πρέπει να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας, τις συμβατικές υποχρεώσεις μας, όπως του ΠΟΕ. δεν μπορούμε να τις παραβιάσουμε αυτές. Ούτε μπορούμε να ανεχθούμε χάριν της καταπολέμησης του dumping παραβιάσεις. Εκτός εάν υπάρξουν διαπιστωθούν στρεβλώσεις στις εξαγωγές. Αν μια χώρα δηλαδή εσκεμμένα παραβιάσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει όπως τα εργασιακά, τότε αυτό είναι dumping ή έμεση επιχορήγηση. Τέλος, η αποτελεσματικότητα των μέτρων είναι το κλειδί και υποστηρίζω την Κομισιόν που ζητάει περισσότερους πόρους για το προσωπικό και για τεχνικά θέματα, για τη λειτουργικά. Γιατί το ίδιο κάνουν και η ΕΠΑ και η Αυστραλία που φροντίζουν τα συμφέροντά τους με σοβαρό τρόπο ως προς τις τον δίκαιο ανταγωνισμό. Σας επανευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι σε λίγο θα υπάρξουν όλα αυτά γραπτός στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. The reason why I